Ο πρώτο θέμα στην ε, σημερινή ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση Κάζα για το μέλλον του ΦΠΑ και δίνω το λόγο στον ομιλητή για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον ε, Επίτροπο. Η έκθεση αυτή αποτελεί ένα, μια βασική διαδικασία η οποία ξεκίνησε το 2010 όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ε, την έκθεση σχετικά με το ΦΠΑ και το σύστημα έχει, ε, περιλαμβάνει πάρα πολλές ε, διοικητικές δαπάνες οι οποίες είναι πολύ ψηλές και επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις. Επίσης ε, όσον αφορά την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ιδίως όταν πρόκειται για συναλλαγές εντός των συνόρων που ε, μπορεί να κοστίζει δισεκατομμύρια δολάρια ε, στους, ε, στα κράτη-μέλη η κατάρτιση αυτή και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια ευρεία διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους. Εγώ συναντήθηκα με πολλές οργανώσεις καθώς επίσης και με εκπροσώπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τώρα θα σας εξηγήσω πού κατέληξα. Ένα από τα πιο βασικά σημεία σε αυτή την έκθεση είναι το γεγονός ότι πρέπει να αντιληφθούμε την υπάρχουσα κατάσταση και να προχωρήσουμε προς τον στόχο μας. Δηλαδή εφόσον πρόκειται για φορολογία μία συναλλαγής η οποία είναι ενδοκινοτική αλλά διασυνοριακή και ε, λαμβάνουμε υπόψη τα στοιχεία που παραβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Πράσινη Βίβλο θεωρούμε δε ότι ε, ε, έχει αποτύχει η πολιτική βούληση μέχρι τούδε και γι' αυτό τώρα πρέπει να βρεθεί μία σωστή λύση και ένα σύστημα μπορεί να είναι αποτελεσματικό μόνο αν συνοδεύει από το σύστημα One Stop Shop και ε, το προβλέπεται αυτή η ρύθμιση από 1η Ιανουαρίου 2015 οπότε ε, θα μειώσει πολύ τα έξοδα ε, για τις ε, διασυνοριακές συναλλαγές στις μικρές επιχειρήσεις. Πρέπει όμως να εξετάσουμε και την πτυχή των συναλλαγών με τρίτες χώρες και ακόμη και αν έχουμε νέα αγορά το πρόβλημα υπάρχει και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αντιμετωπιστεί το ταχύτερο δυνατόν διότι όσον αφορά την ε, καταβολή και την ίσπραξη θα πρέπει να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα και πιστεύω ότι οι καλύτερες μελέτες ήταν ε, αυτές οι οποίες χρησιμοποιούν το πρότυπο αποθήκης και θα πρέπει ε, να αλλάξουμε την υποδομή για να ακολουθήσουμε αυτό το πρότυπο αλλά να προχωρήσουμε πολύ προσεκτικά. Χρειαζόμαστε δηλαδή με περισσότερες μελέτες για να δούμε εάν αυτή η προσέγγιση είναι δεσμευτική. Θα πρέπει ε, να εξετάσουμε όντως τα σημαντικά αυτά θέματα και θα πρέπει ε, να διευκολυνθεί το σύστημα των εξαιρέσεων χρησιμοποιώντας περισσότερο την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ιδίω όσον αφορά τις επιστροφές του ΦΠΑ. Θα σταματήσω εδώ και θα συνεχίσω μετά από τις παρεμβάσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Τον λόγο δίνω τώρα στον Επίτροπο Σεμέτα. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα τον κύριο Κάζα για την θετική και επικοδομητική του έκθεση για την πράσινη βίβλο για την ε, ε, αναμόρφωση του ΦΠΑ διότι νομίζω ότι έχει φτάσει η ώρα να εξετάσουμε ε, το σύστημα ΦΠΑ που ισχύει εδώ και 40 χρόνια. Έχει φτάσει η ώρα λοιπόν να υπάρξει ένα σύγχρονο σύστημα ΦΠΑ που να συνάδει με την ενιαία αγορά και με τα, ε, νέ, τους νέους τρόπους συναλλαγών κατά τρόπον ώστε να συμβάλλει ακόμη καλύτερα μακροπρόθεσμα ή στην ε, ίσφραξη εσόδων. Το σύστημα που παρουσιάστηκε πέρυσι αποτελούσε το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και η σημαντική αντίδραση των ενδιαφερομένων απέδειξε ότι ήταν αναγκαία μια τέτοια, μια ε, τέτοια τέτοια διότι λάβαμε πάρα πολλές ανταποκρίσεις και ε, ουσιαστικά βασιστήκαμε εις ε, τις ε, διαφοροποιήσεις εντός ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πράγμα το οποίο είναι σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιδιαιτέρως και βλέπουμε ότι αναμένονται πολλά από τις μεταρρυθμίσεις αυτής διότι οι αλλαγές του ΦΠΑ απαιτούνται και από τους ενδιαφερόμενους και τις ε, επιχειρήσεις αλλά και ε, τους πολίτες γενικότερα. Θα υπάρξει λοιπόν στη συνέχεια μία ανακοίνωση που θα παρουσιαστεί πρώτου τέλος του έτους για μία συνολική στρατηγική για ε, ένα συνεκτικό σύστημα ΦΠΑ. Δεν θα μπορέσουμε να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα του ΦΠΑ αμέσως αλλά η ανακοίνωση θα αναφέρει αναφέρει τους βασικούς στόχους και ε, θα τονίσει τα σημεία όπου μπορούμε να προχωρήσουμε πιο βραχυπρόθεσμα και που θα χρειαστεί πιο μακροπρόθεσμη εργασία για να έχουμε ε, πιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Και ε, στο πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί για τον επόμενο έτος θα τονίσω μία, έναν από τους στόχους στόχους μας που είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και η σταθεροποίηση. Θα εξετάσουμε τους μηχανισμούς γρήγορης ανταπόκρισης, ε, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ε, και ε, τον τρόπο υποβολής από τις επιχειρήσεις. Κύριοι Ευρωβουλευτές, πολλές φορές στην έκθεση αναφέρονται οι απόψεις των ενδιαφερομένων. Είναι μια φιλόδοξη έκθεση, πράγμα το οποίο είναι ενθαρρυντικό και ε, μπορώ ήδη να σας διαβεβαιώσω ότι θα την εξετάσουμε πάρα πολύ σοβαρά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Επίτροπο και τώρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, Δημοσιονομικού Ελέγχου ο κύριος Στεάζης για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε, συνάδελφε, επίτροπε. Είμαι εισηγητή ε, από πλευρά τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και υπό αυτή την έννοια θα πρέπει να κοιτάξουμε τι μπορούμε να πούμε για τα μέτρα κατά τη απάτη. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο δεν είναι στην αρχή στην έναρξή του. Έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια, είδαμε πριν από κάποια χρόνια την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου που επισήμανε τις ε, αδυναμίες και τα ελαττώματα του συστήματος και βλέπουμε ότι όλα αυτά αποτυπώνονται και στην έκθεση Bowles, στην οποία έκανε αναφορά και ο εισήγητής που περιλαμβάνει πολλές συστάσεις. Ελπίζω οι συστάσεις αυτές περαιτέρω να βρουν εφαρμογή. Το σύστημα, όπως ξέρετε, έχει αδυναμίες και επιτρέπει μαζική απάτη. 80 με 100 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται. Πρόκειται για ένα τεράστιο ποσό για την ε, ε, δημοσιονομική απάτη στην Ευρώπη. Στο σύνολό της υπολογίζεται 200 με 250 ε, δισεκατομμύρια και νομίζω ότι επειδή ο ΦΠΑ αποτελεί μεγάλο τμήμα του ποσού αυτού, αποτελεί ένα μεγάλο κίνητρο για να δράσουμε και μιλάμε για απάτη διασυνοριακή, άρα διασυνοριακά θα πρέπει να είναι και τα μέτρα και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ ε, των κρατών μελών και με την Ευρωπόλ, με την ε, Eurojust, με την Olaf. Και αυτές είναι οι συστάσει ε, τις οποίες απευθύναμε και ω Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους, ε, τον εισηγητή και την Επιτροπή του γιατί ε, συμπεριέλαβαν τις συστάσεις μου όλη την ε, έκθεση μεταξύ των, ε, των παραγράφων 43 και 47. Να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα συμπεριλάβετε στις τάσεις αυτές. Μιλάμε λοιπόν για τη συνοριακή συνεργασία και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και την ευθύνη και τον κίνδυνο που συνεπάγεται τέτοια απάτη στα κρατημέλη. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται και διασυνοριακή και ομοιόμορφη ε, ομοιόμορφο ε, ορισμό σε σχέση με το τι αποτελεί απάτη ως προς τον ΦΠΑ κατά την ε, κατάρτιση της έκθεσής μου. Μίλησα με πάρα πολύ κόσμο, με πολλούς επιθεωρητές και ήταν σαφής, ρητή η επιθυμία τους να υπάρξει ένας ενιαίος ορισμός για το τι αποτελεί απάτη για τον ΦΠΑ και να υπάρχουν και ομοιόμορφες κυρώσεις συζητήσαν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει έκκληση για την απλούστευση του νόμου για την καταπολέμηση της απάτης. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή, η, αυτό το αίτημα. Το είπε και ο εισηγητής σε ό,τι αφορά την απλοποίηση της σχετικής ε, νομοθεσίας και την ενοποίηση της νομοθεσίας. Πολλοί επιθερητές, ελεγκτές που αντιμετωπίζουν καθημερινά τέτοιους εγκληματίες μας λένε ότι κοιτάξτε, πρόκειται για διασυνοριακή απάτη, θα πρέπει να υπάρχει διασυνοριακή συνεργασία και έχουμε και το γλωσσικό ζήτημα γιατί η νομοθεσία για το ΦΠΑ του κάθε κράτους αν δεν ξέρουμε τη γλώσσα, πώς θα την κοιτάξουμε, πώς θα την ερευνήσουμε. Και ένα από τα μία από τις σύμβουλες που μου δίνουν είναι να φροντίσουμε να γίνει μετάφραση σε κάποιες βασικές γλώσσες της νομοθεσίας από το ΦΠΑ σε όλες τις χώρες. Τώρα ποιε θα είναι αυτές οι γλώσσες μπορούμε να το συζητήσουμε για το Eurofis που αποτελεί μια βελγική πρωτοβουλία για την σύσταση ενός δικτύου. Είναι πολύ καλή πρωτοβουλία και νομίζω ότι θα πρέπει να δημιουργήσει επιπρόσθετη αξία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να φροντίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαβιβάζονται και στο Κοινοβούλιο οι σχετικέ εκθέσει που θα προκύπτουν, προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια. Νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία τη έκθεσή μου και η χρήση νέων τεχνολογιών, γιατί μπορούν να μα βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε την απάτη στο ΦΠΑ. Αλλά νομίζω ότι αν οι συστάσει ε, του Επιτροπή, της Επιτροπή Οικονομικών Νομισμάτων και του προπολογισμού λεφτούν υπόψη, θα έχουμε μια ισχυρή θέση ως Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταπολεμήσουμε την απάτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τώρα έχει το λόγο η κυρία Ιβάνοβα από την Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών για δύο λεπτά. Δεν βλέπω την κυρία Ιβάνοβα μέσα στην αίθουσα παρόλα αυτά. Επομένως θα δώσω το λόγο εξ ονόματος της Επιτροπής ε, Μεταφορών και Τουρισμού στον κύριο Φέρμπερ. Δύο λεπτά. Ούτε και ο κύριος Φέρμπερ έχει έλθει. Άρα θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση ε, μεταξύ των πολιτικών ομάδων με πρώτο το ΕΛΚΑ και τον ε, κύριο Παλώνη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η πραγματική υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να συμβαδίζει με μια αποτελεσματική πολιτική στον τομέα του ΦΠΑ. Συμφωνώ απόλυτα με τις γενικές κατευθύνσεις της έκθεσης ΚΑΖΑ. Τονίζει ε, διάφορα κενά που υπάρχουν και προτείνει διαδικασίες ώστε τις δυσκολίες αυτές να τις ξεπεράσουμε. Θα παρακαλέσω όμως την Κομισιό να εργαστεί τάχιστα, διότι ήδη έχουμε καθυστερήσει σημαντικά. Το προσεχές ε, λοιπόν σύστημα ΦΠΑ θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ακρίβεια, να είναι πιο συγκεκριμένο και να έχει σαφείς κανόνες. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν ισχύει. Και αυτό βέβαια γνωρίζουμε ότι θίγει περισσότερο τις επιχειρήσεις ιδίως αυτές που αναπτύσσουν και δραστηριότητα εκτός συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη-μέλη λοιπόν πρέπει να έχουν μια πραγματική πολιτική βούληση για να προχωρήσουμε, αφήνοντας κατά μέρος τους εθνικούς εγωισμούς. Κάτι άλλο σημαντικό, για το οποίο έκανε λόγο και ο κύριος Κάζα, είναι ότι πρέπει να μειώσουμε το γραφειοκρατικό άχθος. Με τον τρόπο αυτό και τα διοικητικά έξοδα θα μειωθούν, και καλύτερα θα εισπράτεται ο ΦΠΑ. Υπάρχει δε το εξή παράδοξο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσει ε, καταβάλουν πολύ περισσότερα σε σχέση με τι μεγάλε. Ε, το διοικητικό του κόστο ε, αναλογικά είναι πολύ υψηλότερο. Και επαναλαμβάνω, ιδίω στον τομέα τη διασυνορική δραστηριότητα. Θα πρέπει βέβαια να υπάρχουν και νομικά ηχέγγυα, πολύ πιο στέρεα νομικά ηχέγγυα για τι επιχειρήσει. Περιμένω λοιπόν να έχουμε νέα μοντέλα, αρμονισμένα από κράτος μέλος σε κράτος μέλος και με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες γιατί είναι το στίχημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, οι μικρομεσαίες. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη μελλοντική στρατηγική για το ΦΠΑ θα ήθελα να σας πω το εξής αγαπητοί συνάδελφοι. Θα πρέπει να φροντίσουμε και την δημοσιονομική εξυγίανση. Είμαστε αυτή τη στιγμή εν μέσω μιας δημοσιονομικής κρίσης. Δεν θα πρέπει να πληρώνουν μόνο οι φτωχότεροι και οι πιο αδύναμοι. Πρέπει να διευρύνουμε, να πληρώνουν οι φορολογούμενοι όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο κόμμα αντικαθιστά τον κύριο Φέρμπερ, εξ ονόματο Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, ή κυρία, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Το πρόβλημα των δημόσιων οικονομικών σε πολλά κράτη-μέλη είναι γνωστό. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το επαναλάβω. Δεν θέλουμε λοιπόν ε, ιδεολογικές ε, μάχες εδώ. Ε, το θέμα είναι πώς θα κάνουμε πιο υγιή και εύρωστα τα δημόσια οικονομικά. Με χαρά διάβασα την έκθεση Κάζα. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά ο συνάδελφος. Η έκθεση του στηρίζεται και στην εξαιρετική πράσινη βίβλο της Κομισιόν, εστιάζει ωστόσο στα σημαντικότερα στοιχεία αυτής. Με εντυπωσίασαν ιδιαίτερα οι ιδέες του σε ό,τι αφορά την περιστολή της απάτης. Ζητείται από τους πολίτες να κάνουν όλο και πιο πολλές θυσίες για να βοηθήσουν ε, την ανάκαμψη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δεν μπορούμε επομένως ε, να αφήσουμε τα πλευρά μας εκτεθειμένα στην απάτη. Από την άλλη πλευρά πρέπει να περιοριστεί η γραφειοκρατία. Και βέβαια όχι σε βάρος ε, επιχειρήσεων που πλήττονται ήδη. Μια άλλη πτυχή η οποία θα πρέπει να τονιστεί και εκεί έχει κάνει πολύ καλές προτάσεις ο κύριος Κάζα. Συγκεκριμένα μια πιο υγεία αν θέλετε, ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς δηλαδή μεγαλύτερη αποδοτικότητα, πιο απλουστευμένες διαδικασίες για τις εταιρείες. Έτσι θα είναι πιο εύκολες οι ε, διασυνορικές συναλλαγές, οι συναλλαγές μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Αυτό μπορούμε όλοι να το υποστήριξουμε, ιδίως σε τέτοιες ε, στιγμές, σε τέτοιες εποχές που πρέπει να δώσουμε κίνητρα στην ε, αγορά, ώστε η Ένωση να αρχίσει να παράγει και πάλι πλούτο. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Κάζ για την έκθεσή του. Είναι άρτια, ισορροπημένη και εστιάζει στι πραγματικέ προτεραιότητε. Είναι καιρό να περάσουμε από τα λόγια στα έργα. Ευχαριστώ. Εγώ σα ευχαριστώ, κύριε Κόμη. Τώρα εκ μέρου ε, των Σοσιαλδημοκρατών, ο κύριο Ελχαντράουι για τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, για να ξεκινήσω θα ήθελα να ευχαριστήσω τον, τον εισηγητή για την εξαιρετική συνεργασία η οποία μας οδήγησε σε μια καλή έκθεση για την οποία να μπορούμε να πούμε ότι σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ στην Ένωση ότι θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική, πιο διαφανής και πιο αποδοτική η διαμορφώσή του και νομίζω ότι η έκθεση του συναδέλφου Κάσα συνεισφέρει, συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή. Αναφέρθηκε ότι βρισκόμαστε σε μια μακρά διαδικασία και αναμένουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να κάνουμε το επόμενο βήμα. Θα πρέπει να διαπιστώσουμε στη συζήτηση ότι τα τελευταία χρόνια έγιναν ε, μετατοπίσεις τα τελευταία χρόνια από ε, άμεσους σε έμεσους φόρους. Αλλά δεν είναι αρκετές αυτές οι αλλαγές για να εγγυηθούν το κράτος εφημερίας. Και γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας ε, σε ό,τι αφορά την ενεργειακή φορολογία την ε, έμεση φορολογία κτλ. Φυσικά ο ΦΠΑ δεν είναι κάτι ουδέτερο, πρόκειται για κάτι το οποίο άμεσα επηρεάζει την καταναλωτική συμπεριφορά του κόσμου. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να ενθαρρύνουμε, να μην ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις. Γι' αυτός λοιπόν ε, θα πρέπει να παραμείνει δυνατότητα μείωση του ΦΠΑ, απαλλαγή από το ΦΠΑ, για παράδειγμα, για συγκεκριμένους λόγους, για κοινωνικούς λόγους και σε κάποιες περιπτώσεις. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης τις νέες εξελίξεις και τις πολιτικές προτεραιότητες, για παράδειγμα, στις μεταφορές, στις μεταφορές και στις ναυτιλιακές μεταφορές υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση από ό,τι στις σιδηροδρομικές ε, μεταφορές. Νομίζω ότι όλα αυτά δυσκολεύουν και μπορεί να προκαλέσουν και στρεβλώσεις και το ίδιο βλέπουμε και στον πολιτισμικό κλάδο όπου όλα τα βιβλία ανεξάρτητα από... θα πρέπει να ε, τη χάνουν τους ίδιες μεταχείρισεις. Θα πρέπει να είναι ίδια η φορολόγηση των βιβλίων σε κάθε περίπτωση εγγράφων ή μη. Τέλος, σε θέματα αποτελεσματικότητας και απάτης, είπαν και άλλοι συνάδελφοι ότι θα πρέπει να μειώσουμε αυτό το τεράστιο ποσό 80 ως 100 δις απόλυες κάθε χρόνο σε ΦΠΑ. Είναι απαράδεκτο αυτό. Χρειάζεται λοιπόν καλύτερη συνεργασία, καλύτερο συντονισμός, καλύτερος έλεγχος. Εμείς ασφαλώς είμαστε υπέρ της απλοποίησης, αλλά υπό τους όρους πάντα ότι δεν θα ανοίξουν παραθυράκια με τον τρόπο αυτό. Και όντως θα καταπολεμηθεί η απάτη στον ΦΠΑ. Υποστηρίζουμε επίσης την αρχή του τόπου κατανάλωσης και αυτό θα πρέπει να συνοδευτεί από την αρχή της μονοθυριδικής αντιμετώπισης στα κράτη-μέλη. Θεωρώ λοιπόν ότι η πρόταση αποτελεί ένα καλό βήμα προς τα μπροστά και αναμένουμε με ανυπομονησία την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει η πρόεδρο. Από του Φιλελεύθερου, ο κύριο Χάκλουντ. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχά τον εισηγητή, ο οποίο πραγματικά κατάρτισε μια πάρα πολύ καλή έκθεση. Να ευχαριστήσω και του κοιόδε εισηγητέ επίσης. Νομίζω ότι εν γέννη η έκθεση είναι πάρα πολύ ποιοτική. Και θα ήθελα τώρα να κοιτάξουμε τις φοροαπαλλαγές σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ και σε ό,τι αφορά τις μη κερδοσκοπικές ε, οργανώσεις. Ε, κάποιοι εξημών ανησυχούμε ιδιαίτερα και μάλιστα ανησυχήσαμε πριν από κάποιους μήνες όταν ήρθατε στο Στρασβούργο και μας επισκεφθήκατε. Θα ήθελα λοιπόν να ταχθώ υπέρ της συνέχισης αυτής της ύπαρξης απαλλαγών για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Θα προσέξετε ότι κι άλλοι συνάδελφοι πέραν μου σχολίασαν και μάλιστα φρόντισαν να επισέλθουν τα σχόλια αυτά στην έκθεση για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι έρχεται όπου να είναι και το Ευρωπαϊκό Έτος για τον εθελοντισμό και αρκετά κράτη-μέλη προβλέπουν τέτοιες απαλλαγές από το ΦΠΑ στα φορολογικά του συστήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως έχει ξεκινήσει διαδικασίες κατά των κρατών μελών αυτών σε κάποιες περιπτώσεις συμπεριλαμβανομένης και της Σουηδίας. Νομίζω ότι είναι μια σαφής πλειοψηφία που έχει δημορφωθεί εδώ στο Κοινοβούλιο η οποία δεν συμφωνεί με την ε, στάση αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ελπίζω να μην συνεχίσουν αυτές οι διαδικασίες. Η έκθεση λοιπόν, όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ καλή και θεωρώ ότι η φοροαπάτη αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει να καταπολεμήσουμε για να αυξήσουμε τα έσοδά μας, ιδιαίτερα στην τρέχουσα κατάσταση. Τέλος, να έχουμε υπόψη μας ότι ο ΦΠΑ αποτελεί ένα σημαντικό κλάδο όπου κινούμαστε προς την κατεύθυνση της ενοποίησης και νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσει αυτό το ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα για την ECR, ε ο κύριος Fox. 1,5 λεπτό. Μπορώ να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή κύριο Κάσα για την εξαιρετική έκθεσή του διότι οποιοδήποτε, οποιαδήποτε έκθεση για την φορολογία είναι αμφιλεγόμενη διότι η φορολογία ε, είναι αρμοδιότης ενός κυριάρχου κράτους και ε, γι' αυτό θέλει ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να έχει τη δυνατότητα δυνατότητα να φορολογεί τους πολίτες μας και η δικιά μας παράταξη δεν το επιθυμεί. Ε, χαιρετίζω όμως τη διατύπωση της εκθέσεως και βλέπω ότι έχουν αφαιρεθεί οι αναφορές στο φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών για να αποφύγουν επιπρόσθετα βάρη στις επιχειρήσεις. Επίσης νέες προτάσεις για το ΦΠΑ θα πρέπει να ε, ε, μπορούν να αμυνθούν κατά της φοροδιαφυγής. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει μια πιο συντονισμένη αντιμετώπιση του ΦΠΑ και αυτό θα αποτελέσει ένα βασικό βήμα για την ε, σωστή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Εκεί που διαφωνώ με την έκθεση αυτή είναι στην παράγραφο 46 όπου ζητάται από τα κράτη-μέλη να αυξήσουν την εναρμόνιση μεταξύ ε, κρατών. Ε, δεν είναι μία πρόταση όμως με την οποία θα συμφωνήσει η πολιτική μου ομάδα διότι ε, μεταξύ του, τα θέματα όπου είναι η φορολόγηση και ο τρόπος φορολόγησης είναι αρμοδιότητα εθνική. Τώρα ο κύριος Χουντής για ένα λεπτό για την ΚΟΕ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεση έχει μέτρα αντιμετώπισης μείωσης της γραφειοκρατίας αλλά δεν διακρίνω όχι τόσο στην έκθεση όσο και στις προθέσεις της κομισιόν την ισχυρή πολιτική βούληση να χτυπηθεί το φαινόμενο των επαγγελματιών φοροφυγάδων η φοροδιαφυγή όσο αφορά το ΦΠΑ αναφέρεται και στην έκθεση είναι 100 δισεκατομμύρια αποκρύβονται και έσοδα από το ΦΠΑ της τάξη του 11%. Η δεύτερη όμως παρατήρηση, η πιο ισχυρή παρατήρηση της ομάδας μας είναι ότι μέσω αυτής της ενίσχυσης παγιώνεται ενδεχομένως η τάση μετακίνησης της φορολογίας από τους άμεσους στους έμεσους φόρους με συνέπεια η πολιτική που ακολουθεί η ευρωπαϊκή ένωση να είναι μείωση των άμεσων φόρων μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων μείωση της φορολογίας των πολυεθνικών αύξηση των εμέσων φόρων του ΦΠΑ στα καταναλωτικά είδη που την πληρώνουν οι μισθωτοί μαζί με τις άλλες περικοπές με συνέπεια να έχουμε ένα άδικο καθεστώς και επομένως το μέλλον του ΦΠΑ με τέτοια χαρακτηριστικά και το μέλλον της φορολογικής πολιτικής να είναι αντίθετο από το μέλλον μιας ευημερούσας οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Τώρα ο κύριος ο, Πάξας για την EFD. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ε, ε, παρουσιάσω ορισμένα σχόλια σχετικά με την έκθεση αυτή διότι το τωρινό ο σύστημα εισπράξεως του ΦΠΑ είναι ένα πεπαλαιωμένο ε, σύστημα και λόγω της κρίσης πρέπει σίγουρα να αντικατασταθεί. Δεύτερον, η αναμόρφωση του ΦΠΑ πρέπει να υπάρξει γρήγορα και να ανταποκριθεί ή στις ανάγκες των καταναλωτών διότι αυτοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα το οποίο να προβλέπει λιγότερο ΦΠΑ σε τομείς που δεν χρειάζεται. Ευχαριστώ και για τους μη εγγεγραμμένους ε, η κυρία Σιανκλέρ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. ΦΠΑ λέγεται ότι είναι ένας φόρος πολυτελείας γιατί είναι πολυτέλεια για αυτούς που μπορούν να τον πληρώσουν. Υπάρχουν συνήθως οι πλούσιοι που αποφεύγουν την καταβολή του και οι φτωχοί μέσω της αγοράς ε, ε, καυσίμων ε, θέρμανσης και βασικών υλικών που τον πληρώνουν. Επιπλέον το ποσό το οποίο καταβάλει το Ηνωμένο Βασίλειο ή ε, την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικό και δεν αναφέρεται από τις κυβερνήσεις ότι δεν πρόκειται για εθνική φορολογία. Πιστεύω λοιπόν ότι η φορολογία αυτή ε, θα έπρεπε να αποφασίζεται όσον αφορά το ποσοστό της από, το κάθε, από την κάθε κυβέρνηση και το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι ο ΦΠΑ στο πετρέλαιο θέρμανσης ε, το οποίο είχε ε, διαταράξει την αξιοπιστία της κυβερνήσεως στη δεκαετία του 80 όταν αυξήθηκε σημαντικά και οι εργατικοί τότε είχαν κατακρίνει την φορολογία αυτή η οποία επεβάρυνε τις ε, φτωχότερες ε, τάξεις αλλά όταν ήρθαν στην αρχή ε, ενέφεραν τη φορολογία αυτή ε, ενώ είχε ζητηθεί να μειωθεί στο 5%. Είναι μια φορολογία η οποία επιβαρύνει τις φτωχότερες τάξεις της χώρας μου και θα έπρεπε να καταργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Τον λόγο τώρα έχει έχουν οι εγγεγραμμένοι ομιλητέ για τις πολιτικές ομάδες. Αν δεν είναι εδώ ο κύριος Χέκμαρ, δίνω το λόγο στον κύριο Δανέλη για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, από οικονομική άποψη ο ΦΠΑ παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία των κρατικών προϋπολογισμών και βεβαίως του ευρωπαϊκού και έτσι με τα γνωστά δημοσιονομικά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό το σύστημα του ΦΠΑ να λειτουργεί τόσο σωστά όσο και αποτελεσματικά. Ως αποτέλεσμα της διοικητικής πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει το υπάρχον σύστημα, το ΦΠΑ δυστυχώς επηρεάζει σημαντικά και τη διοίκηση των επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη. Και ας μην ξεχνάμε ότι υποχρεώσεις όπως η πλήρης ανάκτηση του ΦΠΑ και η ένταξη των διαφόρων πληρωμών του ΦΠΑ στον οικονομικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης είναι πιο εφικτές για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, κάνοντας συγκριτικά δυσκολότερη τη ζωή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δηλαδή του 99% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αφήνουν επίσης και σημαντικά παράθυρα στην απάτη ή τη φοροδιαφυγή. Λαμβάνοντας αυτούς τους παράγοντες υπόψη, οι προτάσεις της παρούσας έκθεσης αποτελούν μια εξαιρετική συνδρομή εκ μέρους του Κοινοβουλίου σε ένα τομέα που δεν υπόκειται στις νομοθετικές αρμοδιότητές του. Μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας, όπως η σύγκληση των γραφειοκρατικών πρακτικών και το ενιαίο ευρωπαϊκό τιμολόγιο, δεν πρόκειται βεβαίως να μεταμορφώσουν το σύστημα του ΦΠΑ, αλλά μπορούν να φέρουν τη διαφορά. Με τα μέτρα σχετικά με τη συλλογή του ΦΠΑ που στοχεύουν στη μείωση της απάτης, τα κράτη-μέλη μπορούν να κερδίσουν μέχρι και δισεκατομμύρια ευρώ και στο θέμα της διασυνοριακής απάτης αν για τη διεξαγωγή αποτελεσματικών ερευνών και τη χρήση νέων τεχνολογιών απαιτηθούν μεγαλύτερες οικονομικές δεσμεύσεις τότε ούτε τα κράτη μέλη ούτε η ευρωπαϊκή ένωση θα πρέπει να τις αποφύγουν. η απλοποίηση δε και η ενιαιοποίηση της νομοθεσίας κατά πολέμηση της απάτης είναι άκρως αναγκαία είναι ευχάριστο πως ε, η έκθεση συνδέει τις μελλοντικές αναθεωρήσεις των συντελεστών και απαλλαγών του ΦΠΑ με κοινωνικές και περιβαλλοντικές προτεραιότητες. Στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών ζητήσαμε μειωμένο ή μηδενικό συντελεστή για τις δημόσιες συγκοινωνίες, το οποίο αν και δεν συμπεριελήφθη στην έκθεση, ελπίζουμε πως θα συμπεριληφθεί στη λίστα αγαθών και υπηρεσιών μειωμένου ΦΠΑ που ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τα κράτη-μέλη. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τη συντονισμένη προσπάθεια που γίνεται για την οδική ασφάλεια με ορίζοντα το 2020, θα ήταν ένα θετικό βήμα αν εποφελούνταν από τη μείωση του ΦΠΑ και τα είδη της οδικής ασφάλειας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σμιτ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά η ομάδα των φιλελευθέρων ε, συνήθω είναι ευνοϊκά ε, διακείμενη, μάλλον στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ευνοϊκά διακείμενη στην πράσινη βίβλο τη Κομισιόν. Σίγουρα θα πρέπει να γίνουν αλλαγέ στο σύστημα ΦΠΑ για να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά. Υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση από τη μια χώρα στην άλλη σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ και αυτό δημιουργεί εμπόδια. Η καλύτερη εναρμόνιση τη πολιτική ε, ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητη για αυτού του λόγου που προανέφερα. Χαιρετίζουμε λοιπόν την περαιτέρω εναρμόνιση των επιπέδων ΦΠΑ. Στηρίζουμε επίση την ιδέα σα ό,τι αφορά την ουδετερότητα του ΦΠΑ. Το υποστηρίζουμε αυτό κύριε Επίτροπε. Θεωρούμε ότι είναι επίση καλή ιδέα και οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις να μην επιβαρυνθούμε επιπρόσθετο φορολογικό βάρος. Ο εισηγητής ξέφρασε και το ενδιαφέρον που θα είχε να εξετάσουμε τις τοπικές και περιφερειακές ε, διαφορετικές συνθήκες και αυτή τη μεταφορά μεταξύ άμεσης και έμεσης ε, φορολογίας. Μπορούμε και πρέπει να μειώσουμε τις εξαιρέσεις γιατί αυτό αυξάνει και το φορολογικό άχθος και την ε, γραφειοκρατία. Μία εξαίρεση βέβαια πρέπει να διατηρηθεί, κατά την άποψή μου, και συγκεκριμένα αυτή αφορά τις ε, οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Έχει ξεκινήσει η Κομισιόν κάποιες διαδικασίες κατά της Σουηδίας που δεν δέχεται την κατάργηση της εξαίρεσης για τους ε, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και αυτό δεν είναι καλό κατά την άποψή μου. Ορισμένοι συνάδελφοι που μίλησαν πριν από εμένα είπαν ότι είναι υπέρ ε, της εξαίρεσης ε, των ε, μικροσκοπικών οργανισμών. Χαίρομαι γιατί υπάρχει υποστήριξη για τις ιδέες αυτές στην Επιτροπή μας, στην Αρμόδια Επιτροπή. Πρέπει να ενθαρρύνουμε το εθελοντικό μη κερδοσκοπικό έργο, άρα δεν θα πρέπει να δημιουργούμε προσκόμματα σε αυτό. Επίσης, θα πρέπει τα ίδια προϊόντα να την χάνουν τις ίδιες αντιμετώπισης σε όλες τις χώρες. Μιλάω για τους ε, φορολογικούς συντελεστές ε, στον τομέα του ΦΠΑ. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον ε, κύριο Κάζα και σας εύχομαι καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας. Η σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στρέιτσεκ έχει το λόγο τώρα για ένα λεπτό. Καλημέρα σας. Ένα λεπτό έχω μόνο στη διάθεσή μου. Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι στο δυνατόν πιο σύντομος και να θέσω τρία σημεία. Το πρώτο, Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε τον κύριο Κάζα. Δεν είναι πολιτικά σωστό, γιατί εγώ σας γνωρίζω, ξέρω ότι είσαστε ε, αφοσιωμένο μέλος ε, του Κοινοβουλίου εδώ και 7 χρόνια ε, στο θέμα του ΦΠΑ και των προβλημάτων του και τουλάχιστον εγώ ξέρω ότι ξέρετε γιατί μιλάτε. Λοιπόν, δεύτερη παρατήρηση. Ο φόβος μου, η ανησυχία μου, μία από τις ανησυχίες μου είναι ότι η στρατηγική του λεγόμενου πράσινου ΦΠΑ, δηλαδή μείωση των συντελεστών για ενεργειακά αποδοτικά φιλοπεριβαλλοντικά προϊόντα και υπηρεσίες, αυτό ίσως οδηγήσει κατά πάσα πιθανότητα σε φοροδιαφυγή απάτες στον τομέα της φορολόγηση. Ε, αυτά δεν μπορούμε να τα αποδεχθούμε, εξού και δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Πέρασε ο χρόνο μου. Ευχαριστώ. Τα υπόλοιπα θα τα πω διμέρως με τον κύριο Κάζα. Μοργάντη τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Κάζα για την καλή δουλειά του και χαίρομαι για την έκθεση όπου αποτυπώνεται το θέμα της ε, διαχείρισης ε, του ΦΠΑ τη μείωση τη γραφειοκρατίας. Έχουμε τα κατάλληλα μέσα στη διάθεσή μα, τα οποία μπορούν να απαλλάξουν το φόρτο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα ήθελα με τον τρόπο αυτό να τονίσω και την τροπολογία μου που ψηφίστηκε σε ό,τι αφορά ένα κατάτατο όριο για το ΦΠΑ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να μειώσουμε το κόστος και να βελτιώσουμε την πρόσβαση στην ενιαία αγορά, ιδιαίτερα για τις νέες επιχειρήσεις. Επίσης γίνονται περαιτέρω προσπάθειες για την περαιτέρω αποτελεσματικότητα της διαμόρφωσης του ΦΠΑ και για να καταπολεμηθούν οι περιπτώσεις κακοδιαχείρισης. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Βέρτμαν, η κυρία Βέρτμαν, ένα λεπτό, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Λόγω της σημασίας του ΦΠΑ ως πηγή εσόδων, για τους προϋπολογισμούς που είναι υποπίεση, κάθε βελτίωση του σημερινού συστήματος είναι επιθυμητή. Και ε, το ΒΠΑ βασίζεται σε νομικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη. Άρα θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τους εφιστάμενους κανόνες. Ε, η πράσινη βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θέλει η πολυπλοκότητα του συστήματος να μειωθεί, γιατί δεν ε, δικαιολογείται για την ενιαία αγορά. Με τα συστήματα ΦΠΑ θα πρέπει να υπάρξει μια ευρεία βάση και αυτό μου φαίνεται λογικό. Οι στόχοι είναι η μεγαλύτερη ε, αποδοτικότητα στη συλλογή των ε, φόρων, οι προσαρμογές στις απαιτήσεις της ενιαίας αγοράς προκειμένου να είναι λειτουργικό το σύστημα συλλογής των φόρων για την διασφάλιση λοιπόν αυτών των εσόδων θα πρέπει να καταπολεμηθούν κατά το δυνατόν οι ε, περιπτώσεις απάτης και ελπίζουμε οι κανόνες να βελτιωθούν προκειμένου η εφαρμογή στα κράτη-μέλη και να είναι χωρίς προβλήματα στο μέλλον και θα ήθελα και να σας ευχαριστήσω εκ νέου για την έκθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Φαϊό, δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση την οποία συζητούμε σήμερα πηγαίνει, θα έλεγα, προς τη σωστή κατεύθυνση. Μας παρουσιάζει μια σύγχρονη εκδοχή για τον ΦΠΑ και τη φορολόγηση εν γέννη και νομίζω ότι διατυπώνει ένα φάσμα προτάσεων που θα πρέπει να ενσωματωθούν στην πρωτοβουλία που θα υποβάλει η Κομισιόν στο Κοινοβούλιο μας. Για όλους αυτούς τους λόγους θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή κύριο Κάζα. Έχω ωστόσο κάποιες διαφορετικές ανησυχίες σε κάποια ζητήματα. Στην έκθεση αναφέρεται η ιδέα ότι ο ΦΠΑ είναι σημαντικό, σημαντική πηγή φορολογικών εσόδων, αλλά ότι επηρεάζει και την λειτουργία της αγοράς πράγματι έχει σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία της ενίας αγοράς. Εξού και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό οι χρήστες να επομίζονται λιγότερο κόστος και λιγότερο διοικητικό βάρος, λιγότερη γραφειοκρατία. Θα πρέπει να καταπολεμηθεί καλύτερα η απάτη και η φοροδιαφυγή. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό τα συστήματα ίσπραξης του ΦΠΑ να βελτιωθούν. Θα ήθελα ωστόσο να τονίσω και το πόσο σημαντικό είναι αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που αυξάνονται οι φόροι, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει και ένα αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών. Ε, από αυτό εξαρτώνται πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πληρώνουν το ΦΠΑ αλλά περιμένουν αιώνες για να ξαναπάρουν πίσω τα ποσά. Και επομένως χρειάζεται ένα σύστημα που θα παρακολουθεί εκ του είναι και στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις ανάγκες τους. Είναι μοχλός ανάπτυξης η ΜΜΕ, μας μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε σε δύσκολους, ταραγμένους καιρούς και θα πρέπει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ληφθούν υπόψη. Το Κοινοβούλιο είναι δεσμευμένο στη βελτίωση του συστήματος ΦΠΑ και αυτό το αποδεικνύει μεταξύ άλλων και η σημερινή έκθεση. Ευχαριστώ, Κορέια Ντεκάμπος, για τρία λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η έκθεση του συναδέλφου Κάζα είναι καλή. Πρώτα απ' όλα, γιατί πρέπει να αναθεωρηθεί ο ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας απαντήσω. Πρέπει να γίνει συμβατό το σύστημα με την εσωτερική αγορά. Όσο περισσότερα είναι τα συστήματα ΦΠΑ, τόσο λιγότερο ευέλικτη είναι και ομαλή η αγορά. Μπορεί να βοηθήσει το ηλεκτρονικό εμπόριο και το εμπόριο γένεια ο ΦΠΑ μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στον κόσμο να επιλέγει τις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών και να μην είναι ένας υποχρεωτικός οφορολογικός συντελεστής. Επίσης θα μειωθεί η φοροδιαφυγή και η απάτη. Μπορούν να γίνουν βελτιώσεις λοιπόν στην ε, αγορά των υπηρεσιών. Επίσης, ε, η ψηφιακή ε, ατζέντα είναι σημαντικό θέμα. Θα πρέπει να δούμε επίσης την τυποποίηση και την υλοποίηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Αυτό λέγεται στο 5, στο 9 μιλάμε για άρση των εμποδίων και φραγμών και αναθεώρηση του συστήματος ΦΠΑ και το ρόλο που παίζει ο ΦΠΑ. Στις ηλεκτρονικές παραγγελίες βιβλίων, για παράδειγμα, και στις κατοίκων πωλήσει. Υπάρχουν θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Το πρώτο είναι η κρίση. Χρειαζόμαστε έσοδα. Χρειαζόμαστε εισόδημα. γιατί νομίζω ότι στα δημόσια ταμεία θα μπαίνουν λιγότεροι φόροι, λιγότερες εισπράξεις λόγω της κρίσης. Άρα ο ΦΠΑ είναι σημαντικό στοιχείο. Επίσης έχουμε προβλήματα δημογραφικά αύξηση του πληθυσμού και στην Ευρώπη. Άρα η γενική τάση είναι η μεταφορά από την άμεση στην έμεση φορολογία. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια νέα ισορροπία μεταξύ άμεση και έμεση φορολόγηση στην Ευρώπη. Τέλο, ε, στο πλαίσιο αυτών των μεταρρυθμίσεων θα πρέπει και η επικουρικότητα να εναρμονιστεί με τι απαιτήσει για την εναρμόνιση. Δηλαδή πρέπει να μειώσουμε το εύρος των συντελεστών ε, ΦΠΑ και να δούμε κατά πόσο θα μπορούσαμε να έχουμε ένα συνεκτικό ε, κατάλογο μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Να ορίσουμε τα κριτήρια, να δούμε τα κατόφλια των εξαιρέσεων της μικρομεσαίας επιχειρήσης. Γνωρίζοντα πάντοτε βέβαια ότι μπορεί αυτές οι εξαιρέσεις να ανοίξουν το δρόμο σε μικρότερη ή μεγαλύτερη κλίμακα φοροδιαφυγή. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Κοζούσνικ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θεωρώ ότι ε, στην έκθεση αυτή ο εισηγητής προσπαθεί να μειώσει το γραφειοκρατικό κόστος ε, και ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν όλο και πιο ηλικιωμένοι υπάλληλοι οι οποίοι ασχολούνται με την επαλήθευση των δηλώσεων του ΦΠΑ και αυτό δημιουργεί επιπρόσθετες επιβαρύνσεις ή στο κράτος και τους πολίτες για να μπορέσουν να ε, προχωρήσουν αυτά τα συστήματα θα πρέπει ε, να ε, μπορέσει να υπάρξει μία μείωση δεν πρέπει να ένιμε να διευρυνθεί η εφαρμογή του ΦΠΑ διότι είναι πολύ δυσμενείς οι επιπτώσεις τους. Ευχαριστώ ότι ο επόμενος ομιλητής δεν είναι εδώ και δίνω το λόγο στον κύριο Στόλογιαν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κρίση οδήγησε πολλά κράτη εις την αύξηση του ποσοστού του ΦΠΑ και άρα το ΦΠΑ είναι μια πολύ, ένα πολύ σημαντικό έσοδο για τα κράτη-μέλη. Κάθε χρόνο λοιπόν μιλώ με τους φοιτητές μου και αναλύουμε τα δίκτυα πληροφοριών και ιδίως αυτό το οποίο δημιουργείται από το ΦΠΑ στην Ευρώπη. Και κάθε φορά οι συζητήσεις με τους φοιτητές είναι πάρα πολύ σημαντικές διότι ότι αυτοί θεωρούν ότι το άχθος του ΦΠΑ είναι πάρα πολύ ε, υψηλό λόγω του ευρωπαϊκού συστήματος που είναι πολύ περίπλοκο Στηρίζω λοιπόν τις συστάσεις του εισηγητή κυρίου Κάζα ο οποίος αποβλέπει εις μία μείωση και κατάργηση στις ε, ε, χώρες μέλη τις απαλλαγές από το ΦΥΠΙΑ οι οποίες απλώς δυσχεραίνουν την γραφειοκρατική εργασία και είμαι βέβαια υπέρ των ε, μέσων που θα μειώσουν τη γραφειοκρατία και ε, θα βελτιώσουν το σύστημα αυτό. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι οι προτάσεις που αναφέρονται εις τις γενικές απαλλαγές για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τις φιλανθρωπικές οργανώσεις είναι καλή ιδέα. Δεν θέλω να δώσω παραδείγματα, αλλά οι περισσότερες από αυτές τις οργανώσεις απλώς συγκαλύπτουν τις δραστηριότητες τους και τα έσοδα που έχουν από αυτές. Ευχαριστώ ο κύριος Λούντιστον για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή είναι καλή και πρέπει να το παραδεχθώ διότι τονίζει τα βασικά θέματα, περισσότερη αποτελεσματικότητα, λιγότερη γραφειοκρατία και λιγότερη φοροδιαφυγή Πρέπει βέβαια να βελτιωθεί η οδηγία αυτή για το ΦΠΑ και πέραν αυτού υπάρχει ένα θέμα που μας απασχολεί σχετικά με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις διότι υπάρχουν αδυναμίες εκεί στην οδηγία και η Δανία, η Αυστρία έχουν κατακρίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι θα ε, να ε, προσαρμόσουν ε, την εθνική τους νομοθεσία σε αυτήν την ευρωπαϊκή ρύθμιση. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουν να υπάρξουν μέσα από την οδηγία εξαιρέσεις για τις ανθρωπιστικές και φιλανθρωπικές οργανώσεις. Περιοριστικά μεν, αλλά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σωστό να δώσουμε ορισμένες δυνατότητες αρμοδιότητες εις, ε, ε, εις οργανώσεις αυτές διότι ε, είναι βασική η δραστηριότητα των φιλανθρωπικών οργανώσεων για την κοινωνία και είναι δυνατόν να υπάρξουν τέτοιες εξαιρέσεις για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Εδώ μιλάμε για φιλανθρωπικά έργα όπως σας είπα που είναι περιορισμένο, που είναι μη κερδοσκοπική, ε, ε, πολλές φορές ε, εκπαιδευτικά ιδρύματα. Άρα δεν θέλουμε να ενισχύσουμε την οικονομική του θέση, αλλά αν ορισμένοι εθελοντικά προσφέρουν τον ελεύθερο χρόνο τους να μην φορολογούνται εφόσον πρόκειται για φιλανθρωπικό ίδρυμα. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να Ξετάσουμε το θέμα των ε, οικονομικών συναλλαγών και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο κύριος Κούρσκι δεν είναι εδώ. Α, τώρα έφτασε η κυρία Κούρσκι και της δίνω το λόγο για ένα λεπτό. Ο κ. Κουρουσκή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι αυξάνοντας ε, τον φορολογικό συντελεστή για το ΦΠΑ στα κράτη-μέλη θα αυξήσει και τα έσοδα του. Αλλά η πραγματικότητα αποδεικνύεται εντελώ διαφορετική και τις τελευταίες 22 ώρες, σύμφωνα με την ε, ε, Ένωση Επιχειρήσεων, σε 22 ε, ώρες μόνο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας θα ξοδέψουν 23.000 ώρες εργασίας για να ασχοληθούμε με τέτοια φορολογικά ζητήματα, γραφειοκρατικά ζητήματα και 20 άτομα θα χάσουν τη δουλειά τους, θα κλείσουν κάποιες επιχειρήσεις. Άρα καλό θα ήταν να υπάρχει ένας ενιαίος φορολογικός συντελεστής για, τους, για τα ίδια προϊόντα και τις ίδιες υπηρεσίες στο ίντερνετ και μη. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι μπορούμε για όλα τα προϊόντα να έχουμε ενιαίο φορολογικό συντελεστή σε όλες τις χώρες. Κάθε χώρα θα πρέπει να αποφασίζει για την φορολογική της πολιτική, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους χαμηλότερους δυνατούς συντελεστές και να εστιαστούμε στην κατανάλωση. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα η κυρία Γκολπέλτς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική του δουλειά, γιατί η οικονομική και η νομισματική πολιτική αποτελούν σημαντικά, σημαντικούς κλάδους και μιλώντας για την ελάχιστη εναρμόνιση. Χωρίς αυτήν δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική η οικονομία της Ευρώπης. Πριν από 40 χρόνια, όταν εισήχθη ο ΦΠΑ, Σκοπός ήταν να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κρατών μελών. Έκτοτε πολλά έχουν αλλάξει και έχουν γίνει διαδικασίες εξυγχρονισμού. Το σύστημα έχει περιπλακεί και πλέον επιβάλλονται στις φορολογικές αρχές και στα άτομα και στους πολίτες υπερβολικά μεγάλα βάρη και αυτό αποτελεί εμπόδιο για την πραγμάτωση της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ε, φοροαπαλλαγή, ε, φοροδιαφυγή, συγγνώμη, φοροαπάτη που ανέρχεται μάλιστα σε ύψος ε, απολειών δισεκατομμυρίων. Επίσης, να διευκρινίσουμε ότι ο ΦΠΑ αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων γιατί μας, βοηθεί, μας βοηθά να χρηματοδοτούμε το σύστημα ευημερίας που έχουμε. Χρειάζονται λοιπόν απαλλαγές, χρειάζονται πλήρεις απαλλαγές. Θα πρέπει να επιτρέπουμε να συνεχίσουν να υπάρχουν αυτές οι απαλλαγές. Δεν θέλουμε να υπάρχουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στο μέλλον. Και εδώ καλωσορίζω πολύ τα μέτρα κατά της απάτης και τα μέτρα απλούστευσης που προτείνει η έκθεση. Εκ παραλλήλου θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη διαφάνειας που υπάρχει. Και αυτό θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος. Επίσης, να κοιτάξουμε και τις διασυνοριακές συναλλαγές, να μην ξεχνάμε και την κατηγορία των συναλλαγών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί προφανώς και αυτές είναι πολύ σημαντικές για την ενιαία αγορά. Έχουν προταθεί διάφορα συστήματα φοροσυλλογής. Νομίζω ότι θα πρέπει να διαλέξουμε κάτι το οποίο τελικά θα αυξήσει τα έσοδά μας. Ευχαριστώ εκ νέου τον γιατί και ευχαριστώ που αποτεχτήκατε και τις τροπολογίες μου. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα ο κύριος Σβάπ, δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, Κύριε Επίτροπε, το σύστημα που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ε, επικρατεί εδώ και 17 χρόνια, αποτελεί για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ένα εμπόδιο σημαντικό σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές τους στην ενιαία αγορά. Είναι περίπλοκοι οι κανονισμοί και είναι διαφορετική η εφαρμογή σε κράτη-μέλη και όλα αυτά οδηγούν σε ένα τεράστιο άχθος, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να συνεχίσουν να δουλεύουν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό διασυνοριακό εμπόριο που έχει τεράστιο δυναμικό ανάπτυξης και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ενιαία αγορά, θα πρέπει να μειωθούν τέτοιου είδους εμπόδια αφορολογικά. Γιατί αυτό ωφελεί στο τέλος και τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Στην τρέχουσα κρίση, η νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πραγματικά απαραίτητη επιτροπή. Και καλωσορίζω και τη συζήτηση για την Πράσινη Βίβλο. Είμαστε υπέρ της απλούστευσης ε, της διαδικασίας και της μείωσης των εμποδίων. Ο φίλος μου και συνάδελφος ε, Κάζα πρότεινε σωστά μέτρα, όπως η εισαγωγή μιας ε, ευρωπαϊκής, ενός ευρωπαϊκού λογιστικού προτύπου ή απλοποίηση της προλογικής δήλωσης. Λυπάμαι ωστόσο ότι συχνά από πλευρά των κρατών μελών δεν υπάρχει σωστή συνεργασία για την εφαρμογή της αρχής προέλευσης σε ό,τι αφορά τι διασυνοριακές συναλλαγές. Κατά το παρελθόν δεν ήταν μόνο τα κράτη-μέλη, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο είχαν τοποθετηθεί για το θέμα αυτό. Και η αρχή αυτή που εφαρμόζονται και που θέλουμε να προτείνουμε δεν είναι ίσως η βέλτιστη, αλλά αποτελεί ένα βήμα προς τα εμπρός. Ε, συνολικά, Πρόεδρε, θέλουμε να υπάρξει κανονισμός και όχι οδηγία για να είναι πιο ομοιόμορφη η εφαρμογή στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράλληλα προκειμένου να δημιουργηθεί ένα, ένα λειτουργικό σύστημα για την ενιαία αγορά στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τώρα Εσάγια, δύο λεπτά. Η κυρία Εσάγια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ, Επίτροπε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή Κάζα για την ισορροπημένη του έκθεση. Είναι σαφής η θέση του Κοινοβουλίου που αποτυπώνεται σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ. Είναι διαφορετικοί οι συντελεστέ ε, ΦΠΑ και είναι διαφορετικά και τα συστήματα φοροαπαλλαγή στα διάφορα κράτη-μέλη και όλα αυτά οδηγούν σε δυσκολίε σε ό,τι αφορά μια εύρυθμα λειτουργούσα εσωτερική αγορά. Χρειάζεται λοιπόν μεταρρύθμιση. Στη μεταρρύθμιση αυτή είναι πολύ σημαντικό να ληφθεί υπόψη και η τρέχουσα κρίση την οποία διανύουμε. Είναι λοιπόν σημαντικό η φοροαπάτη και η φοροδιαφυγή να καταπολεμηθούν. Και εδώ απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φορολογικών υπηρεσιών αρχών και χρειάζεται και μια στρατηγική για την πρόληψη της φοροδιαφυγής. Χρειαζόμαστε όμως παράλληλα και μια πράσινη στρατηγική για το ΦΠΑ η οποία όμως δεν θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα. Εκτός αυτών η γραφειοκρατία που συνδέεται με το ΦΠΑ θα πρέπει να περιοριστεί. Ελπίζουμε επίσης στο νέο σύστημα να αντιμετωπιστεί καλύτερα και το θέμα της, των θέσεων εργασίας, γιατί το αποτέλεσμα σε καμία περίπτωση θα πρέπει μάλλον σε κάθε περίπτωση να οδηγήσει σε μια απλούστευση, σε μια διευκόλυνση της κατάστασης. Θα θέλαμε επίσης τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την κοινωνία των πολιτών. Και ελπίζουμε να πραγματοθεί αυτή η δυνατότητα από τα κράτη-μέλη. Δύο λεπτά ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω συγχαίροντας ε, τους συναδέλφους μου, αλλά όλος ε, ιδιαίτερος τον εισηγητή κύριο Κάζα. Η έκθεση του είναι εξαιρετική εξαιρετικό έργο έχει επιτελέσει. Η εναρμόνιση του συστήματος ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και θα μειώσει την γραφειοκρατία και φυσικά και την απάτη. Επομένως, με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τη λειτουργία της ενίας αγοράς, θα συμβάλλουμε στην μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα της Ευρωζώνης αλλά και συνολικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτό το χρειαζόμαστε ευθύ αμέσω η αύξηση τη ανταγωνιστικότητα. Είναι σημαντικό όπω και η καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή. Γιατί θα μπορούσε να φτάνει και σε 100 δι ε, εσόδων ε, οι φόροι που δεν εισπράττονται. Δηλαδή μιλάμε για το 20% στις περισσότερες χώρες μέλη γιατί είναι μεγάλη πηγή εσόδων, ίσως η κύρια πηγή εσόδων ΦΠΑ σε πολλέ χώρε. Άρα θα πρέπει ε, να φροντίσουμε και το διοικητικό να μειωθεί, να υπάρχει η ουδετερότητα, να βελτιωθεί η νομοθεσία για το ΦΠΑ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι εταιρείε δεν μπορούν πολύ απλά να δεχθούν το επιπλέον διοικητικό άχθος για την έσπραξη του ΦΠΑ, ε, ιδίως ε, μιλώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. πάνω από το 99% των επιχειρήσεων στις, ε, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι συγγνώμη, στην ε, Πορτογαλία είναι μικρομεσαίες και δημιουργούν και το μεγαλύτερο εισόδημα. Οι χώρες οι οποίες παίρνουν εξωτερική βοήθεια, που χρειάζονται εξωτερική βοήθεια, θα πρέπει να ελέγχουν τα έσοδά τους. Έχουν αναγκαστεί να αυξήσουν τους φορολογικούς συνδεστές οι χώρες αυτές. Θα πρέπει να είναι σαφή τα κατόφλια και οι εξαιρέσει. Χρειαζόμαστε αλληλεγγύη. Ευχαριστώ. Ματσόνι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ επικαιρή έκθεση και πολύ καλό και το, κύριο, το έργο του κύριου Κάζα για τον καθορισμό τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση του συστήματο ΦΠΑ. Αυτό ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Νομίζω ότι οι στόχοι είναι ευκταίοι. Εναρμόνιση, διαφάνεια, απλούστευση. Και σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση και τα εργαλεία που προτείνονται, ο κύριος Κάζα πολύ σωστά μας λέει ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι θα πρέπει να προστατευτεί η εθνική αυτονομία. Πλήρης επομένω εφαρμογή της αρχή της επικουρικότητας. Δύο σημαντικά σημεία επί των οποίων πρέπει νομίζω να αναλάβει δράση το συντομότερο δυνατό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρώτον οι εξαιρέσει. Πρέπει το σύστημα να διευκρινιστεί και για τις μη κυβερνητικέ και για του μη οργανισμούς. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει η Κομισιό να έχει υπόψη τη την ανάγκη να γίνει μια ξεκαθά, ένα ξεκαθάρισμα όλων αυτών των ε, εξαιρέσεων που δεν χρησιμοποιείται με σωστό τρόπο και δίκαιο τρόπο. Επίσης, μείωση της γραφειοκρατίας, προσαρμογή του συστήματος, ε, ώστε να ληφθούν υπόψη νέες τεχνολογίες, η καινοτομία. Όλα αυτά είναι σημαντικά και για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και για την ευρωπαϊκή αγορά. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ματσόνη. Τώρα ερχόμαστε στη διαδικασία Catch the Eye. Έχουν ζητήσει το λόγο αρκετοί συνάδελφοι. Ο χρόνο μα επιτρέπει να τον πάρουν το λόγο, αλλά σεβαστούν το ένα λεπτό σα παρακαλώ. Ξεκινάμε από τον κύριο Λούαν. Κύριο Λούχαν για ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ο ΦΠΑ αποτελεί ένα απαραίτητο πόρο για τους εθνικούς προϋπολογισμούς και είναι η βασική του σύσπραξη. Στην αρχή ξεκίνησε με ένα ποσοστό 8% των εσόδων των κρατών μελών και με την αύξηση του ποσοστού του ΦΠΑ αυξήθηκαν και οι εισπράξεις και αντιπροσωπεύονται Αντιπροσωπεύουν όμως 60% των γραφειοκρατικών δαπανών των επιχειρήσεων και γι' αυτό σε μία περίοδο κρίσεως χρειάζονται οικονομίες και θα ήθελα πολύ σύντομα να μπορέσουν να ε, εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις ε, για τις φοροαπαλλαγές από τον ΦΠΑ ε, που δυσχεραίνουν την ζωή των επιχειρήσεων είναι ένα περίπλοκο σύστημα το οποίο επιβαρύνει τη γραφειοκρατία και μειώνει και το ενδιαφέρον της Ευρώπης για το θέμα αυτό. Ένα λεπτό, κύριος Γκούτας, παρακαλώ. Κούτας. Ευχαριστώ πολύ. Κούτας. Ευχαριστώ. Στην ε, κατάσταση αυτή κρίσεως το ΦΠΑ είναι σημαντικός πόρος για τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Η αύξηση αυτή δεν προϋποθέτει οικονομική αύξηση ιδίως όταν ε, πλήττονται τα βασικά προϊόντα και εις ε, τη Ρουμανία παρέμεινε το ποσοστό του ΦΠΑ στο 24% που δεν βοήθησε την κατανάλωση και διαιωνίζει την φτώχεια. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη μας ότι οι καταναλωτές υποφέρουν λόγω της αυξήσεως του ΦΠΑ όπως άλλωστε και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό και χαιρετίζω την πρόταση του εισηγητή να υπάρξει ένα σημείο εκκινήσεως του ΦΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μείωση του κόστους διαχειρήσεως. Κύριος Ρούμπιξ έχει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ εκτιμώ πολύ την εργασία την οποία έγινε για να αναλυθεί η κατάσταση του ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι όλα αυτά τα οποία έχουν αναγραφεί εδώ αποδεικνύουν ότι κατά τα τελευταία 17 χρόνια ε, η ίσπραξη αυτής της φορολογίας είναι ακόμη πιο δύσκολη, πιο κατακαιρματισμένη και δίνει πολλές ε, δυνατότητες για φοροδιαφυγή. Θα πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή ε, να μην πεταλώσουμε ένα ήδη άρρωστο άλογο και να πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα λύσουμε το πρόβλημα. Θα πρέπει να αντικατασταθεί ίσως ο ΦΠΑ με μια φορολογία επί του κύκλου εργασιών, πράγμα το οποίο θα εμποδίσει τη φοροδιαφυγή. Ο κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ο ΦΠΑ είναι μια βασική ίσπραξη για τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά με τις διασυνοριακές συναλλαγές υπάρχει σημαντική φοροδιαφυγή και γι' αυτό πρέπει να βρεθεί μια νέα μέθοδος. Πρόκειται ε, για μια εθνική αρμοδιότητα και γι' αυτό η δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι περιορισμένες. Υπάρχουν όμως ε, ε, πολλές ε, ευκαιρίες για βελτίωση του μηχανισμού, για καλύτερο συντονισμό των εισπράξεων, ιδίως για τις διασυνοριακές συναλλαγές. Θα πρέπει επίσης να μειωθεί το γραφειοκρατικό φορτίο, να γίνονται οι δηλώσεις ΦΠΑ με ψηφιακά μέσα πράγμα το οποίο θα μπορέσει να απλοποιήσει το σύστημα των επιχειρήσεων και να προσφέρει και μεγαλύτερη διαφάνεια. Ευχαριστώ. Την έλλειψη εναρμόνισης ο εισηγητής την ε, επισημαίνει πρόβλημα ή αδυναμία. Εγώ δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Εισπράτεται το ΦΠΑ για την απόκτηση εσόδων ε, και δεύτερο για κάποια οικονομικά αποτελέσματα. Όχι για να φαίνεται ωραίο ο φόρος ή αρμονικός. Κάθε χώρα έχει τη δική της, ε, ε, τις δικές της ανάγκες για την εισπράξη των φόρων. Αυτό πρέπει να ορίζει το φορολογικό σύστημα. Δεν θα πρέπει να εισπράττονται έτσι οι φόροι, ούτε πρέπει να είναι οι ίδιοι με τις διπλανές χώρες. Εγώ θα τον αντικαθιστούσα, αντικαθιστούσα τον ε, ΦΥΠΑΛΦΑ, δεν θα τον ε, εναρμόνιζα. Δεν είναι καλός αυτός ο φόρος, διότι τον ε, πληρώνουν δυσανάλογα άτομα τα οποία δεν έχουν τόσο τις δυνατότητες τον να πληρώνουν. Και θα πρέπει να είναι τελείως διαφορετικό ο τρόπος του, της ίσπραξης και του υπολογισμού. Φοβάμαι όμως ότι οι διατάξεις αυτές θα είναι θύμα της εναρμόνισης ε, και δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να είναι κανονισμός και όχι οδηγία. Εγκέρση. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι εκπρόσωποι ε, κάποιων δάσεων. Ε, λένε συνεχώς τα ίδια σε ό,τι αφορά ε, το ΦΠΑ. Λένε ότι είναι η εναρμόνιση η λύση. Δεν νομίζω όμως ότι ισχύει αυτό. Τι βλέπουμε. Τη Δυτική Ευρώπη. Ποιες δεν βλέπετε πόσο μεγάλες ε, κοινωνικές ανισότητες υπάρχουν και βλέπουμε και πόσο διαφορετικοί είναι οι συντελεστές. Αν συγκρίνουμε Ανατολή και Δύση, θα δείτε πολύ μεγάλε διαφορέ. Στην Ουγγαρία έχουμε ένα επίπεδο ρεκόρ στο ΦΠΑ. 27% θα γίνει. Αυτό προτείνει η Ουγγαρία, η κυβέρνηση τη Ουγγαρία αυτή τη στιγμή. Έτσι θα ξεζουμίσει τον απλό πολίτη. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να παρέμβει πρέπει να παρεμβαίνει όταν έχουμε τέτοια μέτρα τα οποία πραγματικά εξαθλιώνουν τον πολιτή. Θα πρέπει να φροντίσουμε την ευημερία του πολίτη. Η τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Πριν από 40 χρόνια ο φόρος προστιθέμενης αξία εισήχθη και είναι πλέον χρόνο, έχει έρθει πλέον με τον χρόνο να μεταρρυθμίσουμε το σύστημα. Στόχο θα πρέπει να είναι η βελτίωση τη ε, ενιαία αγορά. Η μεταρρύθμιση του συστήματο ΦΠΑ είναι σημαντική για την στρατηγική του 2020 και θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για την ενιαία αγορά, για την ανάπτυξη και για την ενοποίηση των ε, κρατικών προπολογισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε λοιπόν για αυτές τις ε, βελτιώσεις ένα ενιαίο σύστημα ΦΠΑ. Θα πρέπει επίσης ε, να περιορίσουμε, να μειώσουμε τα εμπόδια και το άχθος που βαρύνει τους πολίτες και με τον τρόπο αυτό θα βελτιώσουμε το σύστημα του ΦΠΑ. Το κόστος που συνδέεται με τη συλλογή του ΦΠΑ είναι πολύ σημαντικό και θα μπορούσαμε να τονώσουμε και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων με την απλοποίηση του συστήματος. Είναι σημαντικό να εξευρεθούν λύσεις προκειμένου τα χρήματα να μην καταλήγουν στους αφρολογικούς παραδείσους. Ευχαριστώ πολύ. Ε, άλλοι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, έχει ζητήσει το λόγο και η κυρία Μπασέσκο. Ναι, κυρία Μπασέσκο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον συνάδελφο Κάζα για την έκθεση που πραγματικά είναι εξαιρετική. Τα έσοδα από το ΦΠΑ είναι ένα σημαντικό, μια σημαντική πηγή εσόδων για τους εθνικούς περιπολογισμούς, αλλά σε περίοδο κρίσης καλύτερα θα ήταν να, να, αυξή, να μην ε, έχουμε αύξηση ΦΠΑ και άλλων φόρων. Παραδείγματο χάρη, να σα δώσω ένα παράδειγμα. Στη Ρουμανία ο ΦΠΑ αυξήθηκε κατά 5 ποσοστιαίες μονάδε από το 19% στο 24% και αυτό έχει βλάψει και τον επιχειρηματικό κόσμο και έχει δημιουργήσει πιέσει. Στην αρχή είχαμε πιστέψει ότι είναι ένα τρόπο για να δοθεί νέα όθηση στην οικονομία. Δυστυχώ αυτό το μέτρο καθυστέρησε την έξοδο τη Ρουμανία από την ύφεση. Καλύτερα λοιπόν θα ήταν να είχαμε προχωρήσει σταδιακά σε δύο φάσει. Σήμερα η Ρουμανία είναι ένα από τα κράτη-μέλη με τους ε, υψηλότερους τελεστές ΦΠΑ. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν κίνητρα για την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων αντί να αυξάνουν το ΦΠΑ. Ζήτησε το λόγο και ο κύριος Σκέλη. Έχετε το λόγο κύριε συνάδελφε. Πρόεδρε, για να απαντήσω και στο σχόλιο της συναδέλφου Μπαζέσκου ότι χρειαζόμαστε μέτρα για να τονώσουμε την οικονομία. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι στη χώρα μας ε, η νέα κυβέρνηση έθεσε προτάσεις για να μειωθεί ο ΦΠΑ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στους χώρους εστίασης και αυτό έχει τεράστιο και θετικό αντίκτυπο και για να είμαι δίκαιος για τις πιο πολλές επιχειρήσεις έχει μετακυλιστεί αυτή η απαλλαγή αυτή, η ελάφρυνση και στον καταναλωτή και έτσι έχει βελτιωθεί η κατανάλωση. Άρα σίγουρα υπάρχουν τομείς όπου μπορούμε να τονώσουμε την οικονομία μειώνοντας ε, το ΦΠΑ και η ιδέα να υπάρχει μια, ένας ενιαίος στην Ευρώπη μπορεί να είναι θετικός αλλά δεν είναι ίσως πρακτικά εφαρμόσιμος. Ευχαριστώ. Ε, τελειώσαμε εδώ τις παρεμβάσεις των βουλευτών. Τώρα το λόγο θα πάρει ο Επίτροπος. Ε, Mr. Commissioner, the floor is yours. Uh, thank you, Mrs. President. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές, θέλω να σας ευχαριστήσω και για τα σχόλιά σας και για τις απόψεις που εκφράσατε στη διάρκεια αυτής πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης. Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι ενδιαφερόμενοι φορείς συχνά έχουν κοινέ απόψεις για τις προτεραιότητες και τις δράσεις που θα πρέπει να αναλυφθούν προκειμένου να έχουμε ένα πλούστερο και πιο στεγανό σε σχέση με την ΑΠΑΤ και τη φοροδιαφυγή σύστημα ΦΠΑ στην νέα αγορά. Βλέπω επίσης γενικά ότι στηρίζεται την πρωτοβουλία μας και κάτι, αυτό είναι κάτι ε, πιο απαραίτητο από ποτέ. Θα είναι βέβαια τεράστιο το έργο που μας ε, περιμένει. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι περισσότερες νομοθεσίες βασίζονται στο άρθρο 113 ε, της συνθήκης. Μιλάω για το ΦΠΑ και πρέπει να υπάρξει ομοφωνία στο Συμβούλιο για να εγκριθούν τα μέτρα. Εάν το Συμβούλιο θέλει και αυτό να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες, θα πρέπει να φύγει από το business as usual που φαίνεται ότι το βολεύει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια θα λάβει υπόψη τα συμπεράσματα της προτάσεις, τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα επόμενα βήματα της αναθεώρησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος ΦΠΑ. Όπως σας είπα, ολοκληρώνουμε το έργο μας για την ανακοίνωση σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ σύντομα θα δημοσιευθεί πριν τα τέλη του έτους. Παράλληλα όμως ήδη επεξεργαζόμαστε συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα βελτιώσουμε το σύστημα. Και βέβαια ζητήματα τα οποία σήμερα ε, ακούστηκαν στη συζήτηση, το θέμα της απάτης, του καλύτερου συντονισμού των δραστηριοτήτων, ε, των διασυνορικών ε, δραστηριοτήτων μεταξύ κρατών μελών, τα θέματα των εξαιρέσεων, ε, απαλλαγών δηλαδή κτλ. Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε και όταν εφαρμόσουμε την ε, στρατηγική μας θα διατυπώσουμε συγκεκριμένες προτάσεις για όλα αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα να κλείδι να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά το κοινοβούλιο σας και προσωπικά τον κύριο Κάζα για την ε, υποστήριξη που μας δείχνει και για την επικοδομητική του προσέγγιση. Ευχαριστώ. πολύ κύριε Επίτροπε και το, τη, τη συζήτηση αυτή θα κλείσει ο ίδιος ο εισηγητής, ο κύριος Κάζα. Έχετε το λόγο κύριε εισηγητά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι μίλησαν σήμερα διότι μου έδωσαν ενδείξεις για την ψηφοφορία η οποία θα ακολουθήσει. Ε, υπήρχαν διάφορες λεπτομέρειες που αναφέρονται στην έκθεση για τη μείωση των γραφειοκρατικών ε, ε, φορτίων και που είναι σημαντικά για την οικονομία μας στο τέλος πιστεύω ότι αυτοί οι οποίοι υποφέρουν περισσότερο είναι λόγω της οικονομικής καταστάσεως και δεν θα μπορέσει να υπάρξει βελτίωση χωρίς να αλλάξει το τωρινό σύστημα. Εάν βέβαια ε, εξεταστεί αυτό το οποίο έχει ε, ληφθεί υπόψη θα αληθεί το πρόβλημα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρξουν αριθμοί οι οποίοι θα μπορούν να συγκρίνονται με την είσοδο των στοιχείων, να μιλούμε μόνο για αριθμούς, να μην χρειάζονται μεταφράσεις και γι' αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει ένα εκτενή κωδικοποιημένο κατάλογο των υποχρεώσεων που υπόκεινται σε ΦΠΑ για να μην επιβαρύνουμε τις επιχειρήσεις και να ξέρουν οι επιχειρήσεις ότι υπάρχει ένας εκτενής κατάλογος. Οι επιχειρήσεις μπορούν να προοδεύσουν ε, και ε, έτσι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε και τη φοροδιαφυγή η οποία αναπτύσσεται όταν υπάρχει αστάθεια. Ε, χρειαζόμαστε αν έχουμε βέβαια έναν κανονισμό και όχι οδηγία τότε ε, θα υπάρχει πιο ενιαία ερμηνεία. Θέλω τέλος κυρία Πρόεδρε να ευχαριστήσω όλους αυτούς ε, οι οποίοι συνέβαλαν ε, ευρωβουλευτές, προσωπικό, επιτροπές που συνεργάστηκαν και ελπίζω ότι η έκθεση αυτή θα στηριχθεί σήμερα κατά την ψηφοφορία για να μπορέσουμε να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ. Γάζα. Έληξε εδώ η συζήτηση και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα αργότερα στις 11.30. Τώρα ερχόμαστε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η δήλωση της Επιτροπής με θέμα Αμερικανική πράξη για την απασχόληση. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Θα ξεκινήσουμε με εσάς τη συζήτηση.